Καλησπέρα σας. Μπορούμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με την συνεδρίασή μας σήμερα το απόγευμα. Και αν συμφωνείτε μπορούμε να ξεκινήσουμε με τούτη εδώ τη συνεδρίαση με ανανεωμένο ενδιαφέρον μετά από αυτήν την εβδομάδα διακοπής εορτάζοντας τον Άγιο Σούμαν έτσι όπως τον ε, ε, γιορτάζουμε ε, δυστυχώς βρισκόμαστε με λίγα μέλη έχουν γυρίσει όλοι να δουν τις οικογένειές τους και δεν πρόλαβα να μας ξανάρθουν θα ήθελα λοιπόν να σας ανακοινώσω πως αύριο για την απογευματινή συνεδρίαση δεν θα ξεκινήσουμε στις 2 αλλά στις 3. Έχουμε αυτή τη μικρή αλλαγή για όσους σκοπεύουν να έρθουν, οπότε θα ξεκινήσουμε αύριο το απόγευμα στις 3. Ωραία, εγκρίνεται λοιπόν η ημερήσια διάταξη όσοι έχει και μπορώ να συνεχίσω με το σημείο 3 αυτής Να ξεκινήσουμε λοιπόν με την παρουσίαση μιας μελέτης, μιας εξοδικής ανάλυσης, ε, την οποία ζήτησα εγώ με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ένα ενδιαφέρον που συμμερίζονται όλοι οι συντονιστές και είναι μια εις ανάλυση για τη συμβατότητα των κρατικών ενισχύσεων και της χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ζητήσαμε την ανάλυση αυτή γιατί σε πολλές περιπτώσεις ε, είχαμε αμφιβολίες, προβλήματα ε, και κυρίως σε σχέση με τη χρηματοδότηση κάποιων προγραμμάτων. Τελικά λοιπόν όλα επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο ο γενικό προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιμετωπίζεται ως κάτι πιο περίπλοκο ή ως κρατική ενίσχυση ή υπερεθνική ενίσχυση. Οπότε όλοι ενδιαφερθήκαμε να έχουμε στα χέρια μας μία ανάλυση που θα μας ε, εξηγήσει ακριβώς ποια είναι η κατάσταση. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Φίσερ και αυτή τη στιγμή θα ξεκινήσω δίνοντας το λόγο στον εμπειρογνώμονα που είναι ο καθηγητής Φέδων Νικολαίδης Πολλά κείμενα δικά του έχουμε διαβάσει. Είναι καθηγητής στο Κολέγιο της Ευρώπης και στο Πανεπιστήμιο του Μάστρεχ. Και σίγουρα γνωρίζει πολύ καλά αυτά τα θέματα. Κύριε Νικολαίδη, θα σας δώσουμε το λόγο να μας κάνετε την παρουσίαση. Um, thank Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μια σύντομη απάντηση στην ερώτηση που διατυπώνει ο τίτλος μας είναι «Εξαρτάται». Και όπως εξηγώ στο κείμενό μου, ένα μέτρο για τις κρατικές ενισχύσεις, και αυτό το αναφέρουμε στο κεφάλαιο παριθμών 1, είναι το εάν εκπληρούν τα εξής κριτήρια. Πρώτον, Πρόκειται για πόρους που διαθέτει το κράτος, η δημόσια αρχή, προς μία επιχείρηση. Κρατική πόρη. Λοιπόν, δεύτερον, μεταφορά πόρων που προσφέρουν πλεονέκτημα ότι, που δεν μπορεί υπό τις ε, ομαλές συνθήκες αγοράς να εξασφαλίσει η ίδια η εταιρεία. Τρίτον, πρέπει να είναι επιλεκτικό το μέτρο Δηλαδή χορηγείται σε ορισμένες επιχειρήσεις και όχι σε όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη χώρα ή κάποιου συγκεκριμένου τύπου ή κατηγορίας. Και τέταρτον, το μέτρο αυτό πρέπει να είναι ικανό να επηρεάσει το εμπόριο και να στρεβλώσει τον ανταγωνισμό στην αγορά αυτή. Σορευτικά πρέπει να ισχύουν και τα τέσσερα αυτά κριτήρια για να αποτελέσει κρατική ενίσχυση και άρα δυνάμει του άρθρου 1 107 της ε, συνθήκης για τη Λειτουργία τη Ευρωπαϊκή να έχουμε κρατική ενίσχυση ασύμβατη με την εσωτερική αγορά. Όμως αυτό το μέτρο της ασυμβατότητας δεν είναι απόλυτο, διότι υπάρχουν και εξαιρέσεις ως προς την απαγόρευση. για ορισμένου λόγου. Δηλαδή ότι μερικέ φορέ δεν ακολουθεί αυτόν τον τρόπο λειτουργία η αγορά. Δεν μπορεί να λειτουργήσει ομαλά δηλαδή η αγορά και άρα είναι υποχρεωμένο το κράτο να παρέμβει για να αντιμετωπίσει, να αποκαταστήσει αυτή την ανομαλία στη λειτουργία τη αγορά. Και εδώ έχουμε το κεφάλαιο υπαριθμών 1. Στο δεύτερο κεφάλαιο εστιαζόμαστε στο, στη σημασία του ποιοι είναι οι κρατικοί πόροι το νόημα κρατικών πόρων. Δεν εξηγεί η συνθήκη ποιοι είναι οι κρατικοί πόροι, αλλά ε, έχουμε πληθώρα νομολογίας που έχει σχηματιστεί τα τελευταία 60 χρόνια και που εξετάζει το νόημα των κρατικών πόρων. Στο 171 λοιπόν αναφέρεται ότι προκείται για κρατικές ενισχύσεις που παρέχουν τα κράτη-μέλη ή μέσω κρατικών πόρων. Δηλαδή κάνει μια διάκριση. Η ερμηνεία που έχει δώσει με την ομολογία του Ευρωπαϊκό Δικαστήριο προς το κράτος μέλος αναφέρεται σε οδύποτε δημόσια αρχή, σε οδήποτε επίπεδο της διακυβέρνησης, της κεντρικής, της περιφερειακής αρχής, της ε, τοπικής διακυβέρνησης. Η οδήποτε λοιπόν σώμα ασκεί κρατική εξουσία, δηλαδή εξουσία η οποία είναι στις αρμοδιότητες της κρατικές και καταβάλει από το δικό του προϋπολογισμό πόρους, προβαίνει σε μεταφορά δημοσίων πόρων από κράτος μέλος, με την πρώτη έννοια δηλαδή. Τώρα, οι κρατικοί πόροι η Αυτή στόχο έχει να περιγράψει, να καλύψει κάθε μεταφορά πόρων, με οποιαδήποτε μορφή γίνεται αυτή, από σώμα που δεν συνιστά κρατική αρχή, αλλά ελέγχεται από το κράτος. Χαρακτηριστικά σε αυτή την περίπτωση θα μπορούσαμε να δώσουμε το παράδειγμα μιας επιχείρησης που ανήκει ή ελέγχεται, ε, ανήκει κατά 51% τουλάχιστον ε, των μετοχών της ή ελέγχεται από το κράτος. Φερρυπίν, ε, Υπουργείο των Οικονομικών ή Εμπορίου μπορεί να ορίζει ή να απολύει το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής της επιχείρησης για να είναι κρατική επιχείρηση. Άρα το κράτος έχει καθοριστική επιρροή στις αποφάσεις της επιχείρησης. Πλην όμως το δικαστήριο έχει επίσης σε, αρκετά, ε, σε αρκετές από τις αποφάσεις του επισημάνει ότι δεν αρκεί να ανήκει στο κράτος μια τέτοια επιχείρηση. Γιατί? Διότι έχουν μια δική τους ε, επιχειρηματική ε, ζωή, ένα δικό του επιχειρηματικό βίο αυτέ οι επιχειρήσει ανεξαρτήτω της πολιτική του κράτου. Επομένω, μπορεί να υπάρχει μια τράπεζα η οποία ανήκει στο κράτο και καταρχήν το κράτος μπορεί να υπαγορεύει στην ε, τράπεζα τι πρέπει να κάνει, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι πάντοτε θα ε, συμβαίνει αυτό. Και άρα λέει το δικαστήριο. Επιπλέον του ελέγχου ή της κρατικής διοκτησίας πρέπει είναι απαραίτητο η συγκεκριμένη αυτή απόφαση για τη μεταφορά να ε, υπολογίζεται, να αναγνωρίζεται, να εντοπίζεται ως κρατική απόφαση. Δηλαδή θέλουμε και τον έλεγχο αλλά και την ε, επιβολή μιας απόφασης. Αυτό το εξηγούμε στο δεύτερο κεφάλαιο, το οποίο επίσης αναφέρεται σε μια σειρά από τις κύριες αποφάσεις ε, του Γενικού Δικαστηρίου και του Πρωτοδικίου και μετά πάμε στο τρίτο κεφάλαιο που αναφέρεται στην Ευρωπαϊκή Χρηματοδότηση. Θεωρητικά, τα ευρωπαϊκά κονδύλια πρέπει να παραμένουν εκτός του πεδίου εφαρμογής του 107 διότι το 107 αναφέρεται σε κράτος μέλο ή κρατικού πόρου και δεν αναφέρεται καθόλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν λέει τίποτα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και προφανώς η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι μέλος του εαυτού του. Θα ήταν παράλογο κάτι τέτοιο και ως εκ τούτου αδύνατο. Ωστόσο, επειδή οι περισσότεροι πόροι της Ευρωπαϊκή Ένωση, και θα εξηγήσω ότι εννοώ με το περισσότεροι, όταν διατίθενται σε μια επιχείρηση, όταν χορηγούνται σε μια επιχείρηση, πρέπει να περάσουν μέσα από ένα κρατικό φορέα, ο οποίος επιτοπλίστων είναι μια διαχειριστική αρχή. Και επειδή αυτή η διαχειριστική αρχή έχει τη διακριτική ευχέρεια να επιλέξει την ε, επιλέξιμη επιχείρηση τις επιλέξιμες δράσεις ή τους στόχους για τους οποίους χορηγεί τους πόρους, τότε αυτή η, αυτό το στοιχείο για μένα σωστά θεωρείται ότι αποτελεί και ε, δυνατότητα ελέγχου των πόρων, της διαχείρισης των πόρων, της διάθεσης των πόρων. Στα τα ταμεία παραδείγματι, όπου έχουν τα λειτουργικά προγράμματα τα κράτη-μέλη και τα ελέγχει τα λειτουργικά προγράμματα για να τα εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, χωρί όμω αυτά τα λειτουργικά προγράμματα να ορίζουν κάθε συγκεκριμένη δράση ή να εγκρίνουν τη χορήγηση των πόρων σε κάθε ε, επιμέρους επιχείρηση μπορεί να λάβει οικονομική ενίσχυση μέσα από αυτά τα λειτουργικά προγράμματα. Και επομένως, στην περίπτωση αυτή, έχει σημαντικό βαθμό διακριτικής ευχέρειας το κράτος, η οποία διακριτική ευχέρεια θα επέτρεπε στο κράτος να στρεβλώσει τον ανταγωνισμό. Και ως εκ τούτου ορθώς δίδεται η ερμηνεία ότι ευρωπαϊκοί πόροι που περνούν μέσα από ένα διάβλο που επιτρέπει στο κράτος την άσκηση ελέγχου, μετατρέπει τα κονδύλια σε, ευρωπα... σε εθνικούς, σε κρατικούς πόρους και άρα ε, υπάγει την διάθεσή τους στην ε, περίπτωση του άρθρου 107 των ε, εθνικών ενισχύσεων γιατί επιτρέπει τη στρέβλωση του ανταγωνισμού. Και εδώ λοιπόν έχουμε μια διαφοροποίηση σε σχέση στο 3.1 με τα κονδύλια των οποίων η διαχείριση γίνεται σε επίπεδο κράτους μέλους. Συνοχή επί παραδείγμα, Ταμείο Συνοχής. Μετά περνώ στο σημειο 3.2 στη διαχείριση σε ευρωπαϊκό επίπεδο των κονδυλίων όπου επί παραδείγματι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απευθείας διχειρίζεται ε, ποσά για την έρευνα με το ε, μέσω του προγράμματος COSME ε, ή με άλλους τρόπους. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων διχειρίζεται για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή ιδάλλως τα ποσά πηγαίνουν κατευθείαν στην επιχείρηση χωρίς να διέρχονται από τον διάβλο που θα επέτρεπε στο κράτος μέλος, στον αντίστοιχο φορέα, τον κρατικό, να ασκήσει έλεγχο. Και άρα δεν έχει δυνατότητα κρατικός φορέας με τις αποφάσεις που θα λάβει να προξενήσει στρέβλωση του ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά. Και ως εκ τούτου. Ευρωπαϊκά κονδύλια, των οποίων η διαχείριση γίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο χωρίς να περνούν από τον έλεγχο των κρατών μελών, δεν λογίζονται ως κρατική πόροι που θα υπάγονται στην απαγόρευση ε, του άρθρου 171. Και μακάρι να ήταν τόσο απλά τα πράγματα. Διότι το πρόβλημα, και εδώ ολοκληρώνω προτρέχοντας και κάπως, τη σκέψη μου, γιατί περνάω στα συμπεράσματα πλέον του κειμένου μας, του εγγράφου μας, ε, εδώ έχουμε κανονισμούς πλέον, οι οποίοι αναφέρονται και στην ανάγκη για ε, τα κονδύλια αυτά, τα οποία η διαχείριση γίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τα οποία θα πρέπει να συμμορφώνονται κατά τη διαχείρισή τους με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων. Λογικό αυτό γιατί η συμμόρφωση σημαίνει να μην προξενούν στρέβλωση στον ανταγωνισμό μέσα στην εσωτερική αγορά ανεξαρτήτως το που γίνεται η διαχείριση των ποσών μέσα από τα προγράμματα είτε είναι σε ευρωπαϊκό είτε είναι σε εθνικό επίπεδο στρέβλωση δεν πρέπει να υπάρχει στον ανταγωνισμό, πολύ λογικό. Ωστόσο, εάν μέσα σε ένα κανονισμό διαβάσει κανεί ότι πρέπει να είναι σύμφωνο με του κανόνε περί ε, εθνικών ε, κρατικών ενισχύσεων ή να αποφεύγει την ε, ε, στρέβλωση ή να συμμορφούνται ούτω καθε, ούτω καθεξής, γιατί τέτοιου είδους διατυπώσεις χρησιμοποιούνται, μπορεί να προξενηθεί και σύγχυση. Η συμβατότητα ή η συμμόρφωση προς τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσει. δηλαδή πώς θα, πώς θα ερμηνευθεί. Όταν ζητούμε από τα κράτη-μέλη να συμμορφώνονται με τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις, είναι σαφές το τι εννοούμε. Δηλαδή είτε ακολουθούμε το γενικό κανονισμό απαγόρευσης των κρατικών ενισχύσεων που ε, απαλλάσσει τα κράτη που επιβάλλει ευθέω το 107 για την κοινοποίηση ή αν το μέτρο δεν εμπίπτει στον, στον, στον κανονισμό για τις γενικές εξαιρέσεις τότε πρέπει να γίνεται η κοινοποίηση της ενίσχυσης για, πρώτερη, για προέγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άρα όταν μιλούμε για, κρά... για μέτρα τα οποία έχουν σχεδιάσει και διαχειρίζονται τα κράτη-μέλη είναι σαφές το τι εννοούμε με τη συμμόρφωση. Όταν μιλούμε όμω για ευρωπαϊκά ε, κονδύλια, που, των οποίων η διαχείριση γίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δεν είναι σαφέ τι εννοούμε με τον όρο συμμόρφωση. Ο καθένα θα έχει τη δική του ερμηνεία, εγώ ή ο άλλο, ε, γιατί δεν υπάρχει νομολογία. Αποφυγή των στρεβλώσεων. Ποιο θα αποφεύγει τη στρέβλωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ωραία, πολύ καλά. Βεβαίω και δεν πρέπει να στρεβλώνει τον ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είτε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και Λογικό αυτό. Και μετά πάμε στο κεφάλαιο 3, σε μια ακόμη περίπτωση του σημείου 3-3, που υπάρχει κάτι το ασυνήθιστο. Έχουμε δηλαδή διαρθρωτικά ταμεία που διατίθενται στα κράτη-μέλη και στη συνέχεια αυτά έχουν και τη δυνατότητα, τα κράτη-μέλη δηλαδή, έχουν τη δυνατότητα να τα επιστρέψουν στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων προκειμένου η διαχείριση των κονδυλίων να περάσει μέσα από ένα από τα προγράμματα της ε, ΕΤΕ της ίδιας, της ΕΤΕΠ της ίδιας. Σπάνια συμβαίνει αυτό και μόνο για δημοσιονομικά μέσα. Μάλλον για χρηματοοικονομικά μέσα. Ε, δεν έχουν συγκεκριμένα στοιχεία ποσοστών για το πόσα από αυτά τα χρηματοοικονομικά μέσα επανέρχονται στο ευρωπαϊκό επίπεδο ή πόσα είναι τα κράτη-μέλη που επιλέγουν αυτή την ε, λύση, αλλά μία περιπτωσιολογική παρατήρηση στην οποία έχω, την οποία έχω από την εμπειρία μου συλλέξει αυτή τη στιγμή, μου λέει ότι δύο με τρία κράτη το πολύ πολύ να το έχουν κάνει αυτό. Επομένω, τα τα ταμεία θα μπορούσαν να θεωρηθούν κρατική πόροι. αλλά από το γεγονό και μόνο ότι το κράτο επαναφέρει στο ευρωπαϊκό επίπεδο, στην ΕΤΕΠ, επί παραδείγματι, τα κονδύλια για να τα διαχειριστεί πλέον η ΕΤΕΠ με βάση του δικού τη όρου, το γεγονό και μόνο αυτό οδηγεί στο να θεωρηθούν οι πόροι αυτοί όχι κρατικοί και άρα δεν υπάγονται στους όρους για τις κρατικές ενισχύσεις, αλλά όπως είπα πρόκειται για μία μάλλον ασυνήθιστη σπάνια περίπτωση. Και το τελευταίο τμήμα του τρίτου κεφαλαίου αναφέρεται στην περίπτωση, την νέα περίπτωση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων, έτσι, το λεγόμενο σχέδιο Juncker, στόχος του οποίου είναι ε, να χρησιμοποιεί ευρωπαϊκό χρήμα για να δίνει κίνητρα και για ε, συμμετοχή των ιδιωτών. Δίνει κίνητρα δηλαδή στον ιδιώτη επενδυτή, χωρίς όμως να αποκλείει τη δυνατότητα να συμμετάσχουν και κράτη-μέλη σε μια επένδυση. Αν συμμετέχουν κράτη-μέρη λοιπόν με δικά τους κονδύλια, τότε πρόκειται για κρατικούς πόρους και άρα η ε, διάθεσή τους, η διαχείριση τους πρέπει να ε, συμμορφώνεται με τους όρους για τις κρατικές ενισχύσεις. Και στα συμπεράσματά μου, στο τέταρτο κεφάλαιο, έχω να πω τα εξής. Καρονικά, ευρωπαϊκά κονδύλα, των οποίων η διαχείριση περνάει στα κράτη-μέλη και διοχετεύεται μέσω προγραμμάτων σχεδιασμένων από τα ίδια τα κράτη-μέλη και άρα υπό τον έλεγχο των κρατών μελών, πρέπει να υπάγεται στους κανόνες περικρατικών ενισχύσεων και σε αυτό δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ευρωπαϊκά κονδύλια, των οποίων η διαχείριση γίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, επίσης καταρχήν πρέπει να συμμορφούνται με τις ε, αρχές τις σχετικές με τις κρατικές ενισχύσεις για να αποφεύγουν το, η στρέβλωση της εσωτερικής αγοράς, τον ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά. Άρα κατά κανόνα ή καταρχήν πρέπει να συμμορφούνται με τους κανόνες για τι κρατικέ ενισχύσεις. Η δική μου η θέση είναι ότι ε, όταν ε, υιοθετηθούν και πάλι για την προσεχή περίοδο μετά το 2018 Ήκανος αυτή η αναφορά στις κρατικές ενισχύσεις πρέπει να απαλληφθεί. Δεν χρειάζεται. Διότι ε, ο διαχειριζόμενος ευρωπαϊκό επίπεδο τα ευρωπαϊκά κονδύλια είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και, τα, και οι λοιποί ευρωπαϊκοί φορείς ή θεσμοί δεν πρόκειται αυτοί να προβούν σε στρέβλωση του ανταγωνισμού με στην εσωτερική αγορά. Βεβαίω θα πρέπει να σημειώνεται μέσα στου κανονισμού, αλλά αυτό αρκεί πως δεν πρέπει να οδηγείται σε στρέβλωση ανταγωνισμού η διαχείριση των κονδυλίων αυτών. Άρα καλύπτεται καταρχήν η απέτηση για τι κρατικέ ενισχύσει, αλλά δεν χρειάζεται να αλλάξει τίποτα άλλο, αρκεί να βεβαιούμαστε ότι δεν υπάρχει στρέβλωση του ανταγωνισμού. Ευχαριστώ. Mm, πολύ καλά. Αν όντω ε, αυτό είναι το συμπέρασμα, ε, μετά από όλα αυτά τα τόσο περίπλοκα στοιχεία τα οποία εσείς μας εξηγήσατε και για τη μέγιστη απλούστευση στην οποία αναφέρεστε, μακάρι, μακάρι να τα καταφέρουμε και να γίνει αυτή η προσπάθεια και χαίρομαι πάρα πολύ που κάνατε εσείς αυτή τη μελέτη. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στους συναδέλφους να μας πούν ε, τι πιστεύουν, αλλά επίσης θα δώσω το λόγο και στο Διευθυντή κύριο Κόστρουπ της ε, Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού, γιατί θα ήθελα και αυτός με τη σειρά του να σχολιάσει τα όσα ακούσαμε. Θέλετε να πάρετε το λόγο πριν σχολιάσουν οι συνάδελφοι. Θα ήθελα να σας ακούσουμε εσάς ε, πρώτα. Ευχαριστώ πολύ να σας πω πως λίγα σχόλια έχω να κάνω για την έκθεση. Αυτό που πρέπει να πω είναι ότι αληθεύει και δεν αποτελεί έκπληξη για μένα αυτό. Ο, κύριος, ο καθηγητής κύριος Νικολαίδης είναι πολύ γνωστός, έχει πολύ καλή φήμη στο θέμα αυτό το ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων, οπότε δεν με εκπλήσει που ήταν τόσο ποιοτική η έκθεσή του. Θα ήθελα απλώς πολύ σύντομα να επαναλάβω τα κομβικά στοιχεία για το κατά πόσο κάτι ε, ελέγχεται ως κρατική ενίσχυση ή όχι. Είναι το ποιος αποφασίζει το πώς θα δαπανηθούν τα κονδύλια. Εάν τα κράτη-μέλη αποφασίζουν, τότε ναι, εμπίπτει στον έλεγχο περικρατικών ενισχύσεων. Και αυτό από το 1957 και μετά, γιατί τότε τοποθετήθηκαν στην ε, συνθήκη οι κανόνες αυτοί από την πρώτη και όλα στιγμή. Αν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία αποφασίζει με ποιο τρόπο θα δαπανηθούν τα χρήματα και ποια εταιρεία θα λάβει ποιο ποσό, τότε ναι, δεν εμπίπτει. Όμως, είναι σίγουρα πολύ σημαντικό να αντιμετωπίζουμε τις περιπτώσεις αυτές με συνεκτικό τρόπο και να δούμε και πώς κάνει αυτές τις δαπάνες η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και τι επιτρέπει ως δαπάνες στα κράτη-μέλη. Οπότε οι βασικές αρχές για τον έλεγχο περί ε, κρατικών ενισχύσεων λαμβάνονται υπόψη όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχεδιάζει αυτά τα χρηματοδοτικά προγράμματα και οι βασικές αρχές έχουν να κάνουν με την προσθετικότητα, έτσι ώστε η συμπληρωματικότητα αυτών των κονδυλίων να παροτρύνει επιπλέον επενδύσεις σε σχέση με τις επενδύσεις που θα έχουν σημειωθεί αν δεν παρενέβαινε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Replace private But... και το γεγονό της μη, κυριαρχή της μη υποκατάστασης. Δηλαδή δεν θα πρέπει να υποκαθιστούν τις ε, ιδιωτικέ επενδύσεις αλλά να τις συμπληρώσουν. Αυτές είναι οι βασικές αρχές. Λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό των ευρωπαϊκών προγραμμάτων έτσι ώστε να αποφεύγουμε ε, να στρεβλώνουμε τον ανταγωνισμό. Τώρα για τις συγκεκριμένες συστάσεις που έχουμε στην έκθεση να σας πω πως η Επιτροπή συμφωνεί. Οι κανόνες που εφαρμόζονται θα πρέπει να είναι στο δυνατόν πιο σαφείς και ο καλύτερος τρόπος για να το πετύχουμε αυτό βεβαίως είναι η υποσυζήτηση. Πιστεύω πως οι επόμενες, ε, οι, μάλλον οι προτάσεις που πρόκειται να κατατεθούν στα πλαίσια των επόμενων δημοσιονομικών ε, χρηματοδοτικών προοπτικών θα μας ε, βάλουν στην σωστή κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν κάποιος από τους συναδέλφους που είναι στην αίθουσα θέλουν να σχολιάσουν ή να υποβάλουν κάποια ερώτηση διαφορετικά. Θα ήθελα εγώ να ρωτήσω τον κύριο καθηγητή δύο πράγματα. Στο τελικό σας συμπέρασμα που ζητάτε να μην στευλώνουμε τον ανταγωνισμό και θεωρείτε πως αυτό είναι αρκετό, και θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο ποιο αποφασίζει την ε, δαπάνη ή τη χρηματοδότηση, να σας πω το εξή Πολύ συχνά βρισκόμαστε σε καταστάσεις και πρέπει να σας πω ότι τώρα συζητάμε για πρώτη φορά την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την επόμενη χρηματοδοτική περίοδο. Αυτό που βλέπουμε λοιπόν είναι ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, σε κάποια έργα, έχουμε ένα μείγμα, για να το χαρακτηρίσω έτσι. Δηλαδή, στο ίδιο έργο έχουμε ένα μείγμα. Ε, για παράδειγμα, στα ευρωπαϊκά δίκτυα, όπου έχουμε και αεροδρόμια και κόμβους και λιμένες. Εκεί βρίσκουμε ένα μείγμα χρηματοδότησης και λήψης απόφασης. Δηλαδή, λαμβάνονται κάποιες αποφάσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουμε κάποιους καταλόγους που έχουν υποβάλει ως προτάσεις τα κράτη-μέλη και εκεί οι αποφάσεις επηρεάζουν όντως, δεν θα έλεγα πως τρευλώνουν τον ανταγωνισμό, αλλά σίγουρα επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο οικοδομούνται αυτά τα έργα, δηλαδή πώς συνδέονται, αρθρώνονται αυτά τα έργα μεταξύ τους. Και κάποια κράτη-μέλη, μια και πρόκειται για ευρωπαϊκό διάδρομο ε, και είναι ευρωπαϊκό project, ακόμα και αν όλη η χρηματοδότηση να μην είναι από ευρωπαϊκά κονδύλια, παρόλα αυτά ζητούν ε, κάποιες ε, εξαιρέσεις από τον κανόνα περικρατικών ενεργήσεων. Οπότε, στη δική σας επιχειρηματολογία, τι συμβαίνει με τέτοιες περιπτώσεις, δηλαδή σε τέτοια μεγάλα project που υπάρχει αυτό το μείγμα και υπάρχουν διάφορες εναλλακτικές λύσεις για τη χρηματοδότηση και διάφορες πηγές χρηματοδότησης. Αυτή η απλούστευση, η απλοποίηση που προτείνατε εσείς, έτσι ώστε να μην στρεβλώνουν τα ευρωπαϊκά κονδύλια τον ανταγωνισμό. Πώς μπορούμε να παρακολουθούμε ότι εφαρμόζονται. Ποιοι θα είναι οι όροι που τους οποίου θα κάνουμε αυτή την παρακολούθηση, αυτή την εποπτεία, έτσι ώστε να μην έχουμε στρέβλωση τη στιγμή της χρηματοδότησης, όταν μιλάμε για τόσο μεγάλα project. Η ερώτηση που κάνετε είναι πολύ δύσκολη. Υπάρχουν ε, πολλές ε, πτυχές αλλεπάλληλες μέσα στην ερώτησή σας. Όντως, τα έργα τα οποία είναι παρόμοια στα κράτη-μέλη είναι ανταγωνιστικά μεταξύ τους. Όταν το κράτος μέλος αποφασίζει από μόνο του, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εφαρμόζει τη λογική της κρατικής επιδότησης σε ό,τι αφορά την χρηματοδότηση του έργου και θα λύσει τα αρνητικά με τα σε ό,τι αφορά δηλαδή την κρατική ενίσχυση και τη στρέβλωση του ανταγωνισμού. Όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλείται να αποφασίσει από ένα κατάλογο έργων ποιο θα χρηματοδοτήσει, για παράδειγμα σε έργα στον τομέα των μεταφορών, εκεί πάλι θα πρέπει να ακολουθεί την ίδια λογική. Ποια είναι τα ωφέλη λοιπόν για την Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό τη αποτελεί προτεραιότητα το έργο του εκάστοτε. Το έργο καλύπτει ένα χάσμα, ένα κενό στο πλαίσιο του εφιστάμενο και να τα ζυγίσει αυτά έναντι της ρεύλωσης που θα προκληθεί στον κοινωτικό ανταγωνισμό. Είτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρηματοδοτεί και αποφασίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή είτε αποφασίζει και χρηματοδοτεί το κράτος μέλος, ουσιαστικά η σκέψη από πίσω θα πρέπει να είναι η ίδια. Τα ωφέλη θα είναι πιο πολλά από ότι οι αρνητικέ επιπτώσει, από ότι τη στρέβλωση. Προφανώ, όταν ε, πρόκειται για ένα έργο χρηματοδοτούμενο από το κράτο μέλος, πιο πολύ θα απασχολεί να υπάρχουν ωφέλη για το ίδιο το κράτος μέλος και όχι τόσο πολύ για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα υπάρχει συμπληρωματικότητα, υπάρχει και ενδεχόμενη σύγκρουση. Αλλά παράλληλα υπάρχει συμπληρωματικότητα και μεταξύ των έργων τα οποία σχεδιάζονται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα οποία έχουν σχεδιαστεί για να ωφελήσουν το σύνολο της Ευρώπης. Και αυτών που αποφασίζονται σε επίπεδο κράτους μέλους, η λογική θα πρέπει να είναι η ίδια. Η κατανομή τώρα του ωφέλους δεν ε, είναι η ίδια απαραίτητα στα ευρωπαϊκά και τα εθνικά έργα. Αλλά γι' αυτό υπάρχει αυτή η χρηματοδότηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, υποθέτω, για να υπάρχει μια παραπάνω αξία και να μην λαμβάνονται πάντα αποφάσεις βάσει των εθνικών συμφερόντων. Μπορεί να έχω υπεραπλουστεύσει λίγο την κατάσταση Ομολογουμένως, η εντελεχής αξιολόγηση των έργων αυτών είναι πολύ δύσκολη, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για μακροπρόθεσμα έργα. Και δεν είμαστε πάντα απόλυτα ορθοί. Έχουμε διάφορα παραδείγματα, όπου τα κρατημέλη σχεδιάζουν μεγάλα έργα, αερολιμένες, λιμένες ε, και Ξέρουμε ότι επειδή τα σχέδια αυτά έχουν γίνει από μία και μόνο αρχή, ενδεχομένως ε, μακροπρόθεσμα το ένα να αποδυναμώνει το άλλο. Αυτό δεν είναι μυστικό. Το ελεκτικό συνέδριο, άλλωστε σε μία σειρά ειδικών αναφορών και εκθέσεων, έχει επισημάνει ότι αν δεν υπάρχει μια ολοκληρωτική προσέγγιση όλων των έργων αυτών, που σχεδιάζονται και εφαρμόζονται και υλοποιούνται σε κάθε κράτος μέλος δεν ε, μεγιστοποιούμε όλο το δυναμικό της αξίας που θα είχε ενδεχομένως αυτό το έργο. Αυτό φυσικά είναι θέμα συντονισμού. Έτσι πιστεύω. Δεν τίθεται τόσο πολύ θέμα σύγκρουσης των όσων κάνουν τα κρατη με αυτά που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. δημιουργείται το κόνσεπτ του, του ευρωπαϊκού ε, κοινού συμφέροντος ή ε, το βλέπετε εσείς κάθε φορά κατά... Τα έργα τα οποία χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, α, για τα οποία ε, τα κονδύλια χορηγούνται μέσω των ε, εθνικών αρχών. Thank you. I want to make a distinction. Ναι, αναφερόμαστε στη σύγχυση η οποία προκαλείται σε ό,τι αφορά την αναφορά στη συμμόρφωση με του όρου για την κρατική επιδότηση. Στα σχολεία σα νομίζω ότι αναφέρεται να έχει εξετάσει τον αντίκτυπο στον ανταγωνισμό της ε, χρηματοδότησης ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ενδεχομένω να υπάρχει. Εγώ όμω δεν είμαι τι μελέτε από το λευκό συνέδριο. Αυτέ οι μελέτε αφορούν βασικά έργα υποδομών. Εδώ ο ανταγωνισμός έχει πολύ πιο αρνητικές επιπτώσεις γιατί ο ανταγωνισμός, ο υποδομές, συγγνώμη, ενδεχομένως να χρηστευτούν ε, αν υπάρξει τη χρηματοδότηση έρευνας ή την χρηματοδότηση επιχειρήσεων. Εκεί πιστεύω ότι είναι πιο υγιής ο ανταγωνισμός. Είναι καλό να ανταγωνίζονται διάφορες εταιρείε για τα ίδια κονδύλια, γιατί σε τελική ανάλυση θα κερδίσει το καλύτερο έργο, το οποίο και θα έχει πιο πολλά ωφέλη για την Ευρώπη στο σύνολό τη. Άρα, υπό την έννοια, πιο πολύ με ανησυχούν οι πόροι οι οποίοι δαπανώνται για ανταγωνιστικές υποδομές γιατί εκεί τίθεται θέμα επικάλυψης και απώλειας ουσιαστικά το κονδυλίων. Να κάνω λοιπόν αυτή τη συγκεκριμένη, τη συγκεκριμένη διάκριση ε, της τρέβλωσης που προκαλείται λόγω της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης είναι δύο διαφορετικές υποθέσεις όμως αυτές. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Δεν ξέρω αν κάποιο συνάδελφο θέλει να απαντήσει διαφορετικά. Θα ζητούσα από το διευθυντή ε, της DG Competition να απαντήσει σε όλα αυτά τα επιχειρήματα και στι διαφορετικέ δομέ τις οποίες εμείς πολλέ φορές συναντάμε και στη διαφορετική εφαρμογή που γίνεται ε, όπου έχουμε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση μέσω ταμείων και παράλληλα έχουμε και προτάσεις από τα ίδια τα κράτη-μέλη που ζητούν τμήματα κάποιων project να χρηματοδοτηθούν ως αποκρατικά κονδύλια λόγω ε, δημοσίου Πως πολλές φορές βρίσκουμε τέτοιου είδους project με πολλαπλές πηγές χρηματοδότησης και εκεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι αρχές που εφαρμόζουμε είναι παρόμοιες με αυτές που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν επιλέγει ε, έργα στα πλαίσια του Connecting Europe ή του TEN-T. Οπότε εδώ αντιμετωπίζουμε θέματα όπως η διαφάνεια, τα ξεκαθαρά κριτήρια τα οποία θα πρέπει πριν την επιλογή να έχουν ε, διατυπωθεί, τις, κατά πόσο είναι ε, υπέρ του γενικού συμφέροντος τα έργα αυτά, ε, το κατά πόσο κανόνες ανεξάρτητα με το ποια είναι η πηγή της χρηματοδότησης. Οπότε, οι αρχές που ακολουθούμε ε, για τον έλεγχο των κρατικών για κάθε ευρώ το οποίο ε, δίνουμε εμείς σε μια οικονομική δραστηριότητα ή εμπορική δράση επηρεάζουμε τον ανταγωνισμό και θα πρέπει να περιορίζονται αυτές οι συνέπειες και να είναι μεγαλύτερα τα ωφέλη. Ε, του ίδιου του έργου. Και νομίζω ότι αυτή είναι η αντιμετώπιση που ακολουθούμε και στα μεγάλα και περίπλοκα έργα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξή. Έχουμε και κάποιες περιπτώσεις με κυβερνήσεις οι οποίες λαμβάνουν αποφάσεις για το κατά πόσο σε ένα έργο υποδομής για παράδειγμα Και μιλάμε εδώ πάντα για το εθνικό σκέλος του έργου και την εθνική χρηματοδότηση. Για παράδειγμα για το Connecting ε, Europe ε, ή για, τα, για ε, τη χρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ. Οπότε αυτή η χρηματοδότηση είναι δική σας αρμοδιότητα. Μα του project μπορεί να χρηματοδοτηθεί από εθνικά κονδύλια ε, και κάποιο άλλο κομμάτι μπορεί να έχει ευρωπαϊκή χρηματοδότηση ή ακόμα και να υπάρχει ε, ανταγωνισμός μεταξύ έργων. Τι λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ελέγχει το κατά πόσο έργων και κάποια μένουν εκτός. Κάποια χρηματοδοτούνται μέσω εθνικών κονδυλίων και εμπίπτουν στις ε, ε, διατάξεις περί κρατικών ενισχύσεων και κάποια άλλα χρηματοδοτούνται ε, μέσω ευρωπαϊκών ταμείων. Οπότε τι κάνουν με διαφορετικό τρόπο. Κάνετε κάποιες διαπραγματεύσεις με τα κράτη-μέλη για την κατανόμη της χρηματοδότησης. Γιατί βέβαια οι αποφάσεις αυτές επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό το τι γίνεται επί τόπου. Ναι. Νομίζω ότι αυτός ακριβώς είναι ο ρόλος μας. Μας ανησυχεί λιγότερο το θέμα των μέτρων που λαμβάνουν, ε, τα μέτρα που λαμβάνουν τα κράτη-μέλη. Ανάλυσης, έγγραφο ουσιαστικά καθοδήγησης σε ό,τι αφορά τα έργα υποδομών. Έχουμε για παράδειγμα ένα σημείωμα για το φάσμα όπου προσπαθούμε να εξηγήσουμε στα κράτη-μέλη και σε όποιον ενδιαφέρεται το πώς ισχύουν οι κανόνες κρατικής ενίσχυση για τον εκάστοτε τομέα. Κατά πόσον, θα... Κατά πόσον ε, πρόκειται σε κάποιους ε, κανόνες εξαίρεσης και ποια είναι τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται. Και εδώ φυσικά ο διαστοριακός χαρακτήρας έχει σημαντική επίπτωση. Για παράδειγμα, κοιτάμε, γιατί αυτό θα προκαλούσε προφανώς μεγαλύτερο ανταγωνισμό από ότι σε περιοχές που δεν υπάρχει άλλο αεροδρόμιο. Και φυσικά αν δεν υπάρχει αεροδρόμιο, το όφελος του καινούργιου αεροδρομίου ήταν πολύ μεγαλύτερο για ρίζουν τους κανόνες και να τους λάβουν υπόψη στη φάση του σχεδιασμού ήδη και να ξέρουν υπό ποιου όρου. Σε λιγότερο από ένα χρόνο θα έχει φύγει το Ηνωμένο Βασίλειο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γνωρίζουμε πω στο μέλλον η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να εστιάζει περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν. Πιστεύετε στα όσα συζητάμε μπορούμε να συνεχίζουμε όπως κάναμε στο παρελθόν ή αυτές οι νέες προκλήσεις ε, να αλλάξουμε την ε, πορεία και την αντιμετώπιση που ακολουθούμε. Πολύ φοβάμαι ότι αυτή η ερώτηση ξεπερνάει λίγο το δικό μου τομέα και τις δικές μου αρμοδιότητες. Είναι πολιτική αυτή η ερώτηση. Και πριν από μερικές... Δεν υπάρχει δεύτερο θέμα κρατικού ελέγχου, όταν μιλάμε για άσυλο, όταν μιλάμε για τη μετανάστευση, για θέματα ασφάλειας, όλοι αυτοί οι τομείς είναι τομείς μη οικονομικής φύσης. Άρα, ό,τι ενίσχυση χορηγείται προς τις δραστηριότητε αυτές είτε από τον κινητικό προπολογισμό είτε από του εθνικούς προπολογισμού δεν εμπίπτει στον τομέα των ε, αρμοδιότητων μα, Δεν τίθεται θέμα αρμοδιότητα. Για την ψηφιοποίηση, ναι, υπάρχει αρμοδιότητα. Αν, για παράδειγμα, τα κράτη-μέλη αποφασίσουν να υποστηρίξουν την χύψη εταιρεία και να επενδύσουν σε ναι, παράγουν τέτοια τεχνολογία. Και αν τα κράτη-μέλη επιλέξουν μία εταιρεία να ενισχύσουν για έρευνα η οποία γίνεται μία διάκριση σε ό,τι αφορά τους τομείς που ήδη εξυπηρετούνται και από, μεταξύ των τομέων που δεν υπάρχει. Ναι, ο καθηγητής έχει το λόγο. In my experience. Από την εμπειρία μου. Θα υπερασπιστώ την Επιτροπή, αν και δεν το χρειάζεται. Προφανώ είναι πολύ τόσο να υπερευσεί τον εαυτό τη. Αλλά αν δεχτείτε και τη δική μου τη θέση ω ε, έκφραση ανεξάρτητης φωνής, δεν μου είχε τυχεί ποτέ να έχουν, να έχουν παραβιάσει τα συμφέροντα κράτους μέλους ε, κανόνες ε, κρατικών ενισχύσεων που έχουν παραβιαστεί. Είναι απλά τα ζητήματα που πρέπει να κρυθούν. Δηλαδή είναι λογικό με βάση τους ε, κανόνες της οικονομικής δραστηριότητας, φέρνουν κάποιο πλεονέκτημα, προσφέρονται αυτές οι ενισχύσεις κάπου που μπορούν να βελτιώσουν αποτέλεσμα, υπάρχει ανάγκη παρέμβασης δηλαδή και αν η απάντηση είναι θετική τότε πολύ συχνά πιστεύω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για να μην πω πάντα, θα δώσει καταβατική, καταφατική απάντηση, άρα θα επιτρέπεται η κρατική ενίσχυση. Είναι πολλές οι περιπτώσεις, όπως είπα, δεν έχω δει ποτέ μου το αντίθετο, που έχουν τα κράτη-μέλη θεωρήσει ότι τους περιορίζουν οι κανόνες περικρατικών ενισχύσεων, τους βάζουν σε ένα κορσέ στενό, αλλά δεν έχω δει ποτέ να... Νομίζω πως ε, Εδώ θα ήθελα να ρωτήσω τον διευθυντή της DigiComp εν ώψη και των νέων χρηματοδοτικών προοπτικών και των όσων έχουν γίνει για τα αιτήματα των δικαιούχων αυτών των ενισχύσεων που δεν είναι μόνο κράτη-μέλη για την απλούστευση αυτή ε, της εφαρμογής των κανόνων λαμβάνοντας υπόψη και όλες τις επιπλοκές που θα έχουμε στα προγράμματα λόγω των μειώσεων που θα υποστούν ωστούν αυτοί είναι οι κανόνες και τι συνέπειες θα έχουν όχι μόνο στα τομεακά προγράμματα, αλλά και πιο γενικά. Στις αποφάσεις που θα πρέπει να λάβουμε, ε, πώς θα επηρεαστούμε, γιατί βέβαια θα πρέπει να επιλέξουμε συγκεκριμένες γραμμές του προεκλογισμού, συγκεκριμένα προγράμματα, οπότε είναι υψηλότερο ή θα είμαστε πιο απαιτητικοί, πιο αυστηροί, ακριβώς για να είμαστε σίγουροι πως κανείς δεν θα περάσει ε, μέσα από το δίκτυ αν, ε, μέσα από το δίκτυ, αν δεν το αξίζει. Εσείς τι νομίζετε. Well, I think it's a bit... Νομίζω τις προτάσεις για τα διάφορα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις 18 Απριλίου όμως αν δεν με απατάει η μνήμη μου ε, η Επίτροπος μου, η Επίτροπος Φεστάγερ ήταν εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, για την ετήσια έκθεση ανταγωνισμού αν δεν απατώμε και εκεί ήδη επισήμανε πώς βρίσκονται, εμποδίζουν οι κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις. Και βέβαια να υπάρχει επάρκεια με βάση και άλλους κανόνες ενός ε, ελέγχου υπείου εκεί όπου μιλούμε κυρίως για συνδυασμό κρατικών κονδυλίων και κονδυλίων που προέρχονται από κράτη-μέλη. Αλλά αφού ακόμα είναι να εξηγήσει... Για να το κλείσουμε και δεν ξέρω αν ο κύριος καθηγητής θέλει να μας κάνει κάποια σύσταση σε αυτή τη συζήτηση η οποία ανοίγει αυτή τη στιγμή. Είναι μόνο η προσωπική μου προτίμηση. Δεν νομίζω πως είστε και ο μόνος. Αλλά νομίζω ότι από αυτά που ακούμε, μάλλον προς την αντίθετη κατεύθυνση θα πάμε. Καταλαβαίνω βέβαια πως η δική σας εμπειρία και η δική μας μας οδηγεί σε μεγαλύτερη αυστηρότητα. Εν πάση περιπτώσει νομίζω πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα κάνει τη δουλειά της καλά ό,τι και να συμβεί. Αν συμφωνείτε λοιπόν και δεν υπάρχει κανείς άλλος που να ζητά το λόγο θα μπορούσαμε να περάσουμε στο επόμενο, αφού ευχαριστήσουμε και τον κύριο καθηγητή αλλά και, τον και το διευθυντή της DigiComp που μας έκανε την τιμή να είναι εδώ για τη συζήτηση αυτή. Βρισκόμαστε ακόμα στην αρχή της όλης διαδικασίας, δεν ξέρουμε του χρόνου πώς θα ε, συζητηθεί το θέμα της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης, αλλά υπάρχουν κάποια σημεία στα οποία εμείς Χρειαζόμαστε διευκρινήσεις. Υπάρχουν κάποιες ε, ε, γκρίζες ζώνες ε, και γι' αυτό σας ευχαριστώ πολύ για τη βοήθειά σας. Θα συνεχίσουμε, θα είμαστε σε επαφή και σίγουρα θα συναντηθούμε και κάποια επόμενη φορά. Στις 25 μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος, έχουμε ε, μία ακόμα συνάντηση. Τώρα επιτρέψτε μου να περάσουμε στο επόμενο ε, σημείο της σημερινής διάταξης που είναι η μελέτη σχετικά με τη διασφάλιση της δημιουργίας θέσεων εργασίας υψηλής ποιότητας από τα χρηματοδοτικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πώς μετά τις ακροάσεις που κάναμε και τις μελέτες που έχουμε λάβει, πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε πως προγράμματα όπως το Horizon 2020 θα δώσει καλύτερα αποτελέσματα και θα ενσωματώσει ε, θετικά στοιχεία ε, σε επίπεδο απασχολησιμότητα θέσεων εργασίας, ε, γιατί υπάρχουν κάποια προγράμματα τα οποία έχουμε εντοπίσει και τα οποία ως στόχο είχαν τη δημιουργία απασχόλησης ή τη διευκόλυνση ε, της επιστροφής στην απασχόληση και παρόλα αυτά ε, η επιτυχία τους δεν είναι τόσο μεγάλη και μάλιστα και οι δικαιούχοι δεν έχουν αντιληφθεί τα εκτιματά τους. Έχουμε τις διάφορες πρακτικές που είχαμε στην, στο Horizon 2020 και από τα οποία χρειάζεται να διδαχθούμε ε, ποιες είναι οι σωστότερες πρακτικές. Έχουμε κοντά μας τους συντάκτες της μελέτης την έχουμε μοιράσει Νομίζω λοιπόν πως μπορούμε τώρα να δώσουμε το λόγο στην κυρία Χόφμαν για να κάνει την παρουσίαση. Έχετε το λόγο. Thank you very much. Um, για την έρευνα σε ό,τι αφορά τις πολιτικές και έχω διάφορους συναδέλφους μου εδώ σήμερα και έχουμε όλοι μαζί συνεργαστεί για να εξασφαλίσουμε τη δημιουργία σωστών θέσεων εργασία από την κοινωτική χρηματοδότηση και θα ήθελαμε να σα ε, παρουσιάσουμε κάποια βασικά πορίσματα και συμπεράσματα και πωλήσει και ποιοτικέ ε, θέσει εργασία είναι βασικό στοιχείο τη στρατηγική για το 2020 τη Ευρώπη, προκειμένου να υπάρχει σωστή και ανάπτυξη που θα περιλαμβάνει όλους ε, τους τομείς και όλους τους πολίτες. Δεν γνωρίζουμε πολλά για το πώς... Ε, γιατί πολλοί α, μας ε, ρωτούν πώς ε, είναι η απόδοση των κοινωνικών αυτών πόρων για τη δημιουργία θέσεων απασχόληση υψηλή ποιότητα. Στόχου είχαμε τρει στην μελέτη μα. Καταρχά, θέλαμε να αναλύσουμε τα τέσσερα επιλεγμένα τα σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα δημιουργία θέσεων απασχόλησης υψηλής ποιότητας. Εδώ τονίζω το δυναμικό σε ό,τι αφορά δηλαδή την ικανότητα που έχει το καφεταμείο είναι διαφορετική. Πολύ διαφορετική. Επίσης, κοιτάξαμε πώς τα πήγε το καφεταμείο. Το πώς μετράτε η δημιουργία θέσεων απασχόλησης και η ποιότητα θέσεων απασχόλησης στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης. Και τρίτον, είχαμε ως στόχο να εντοπίσουμε κάποια βασικά χαρακτηριστικά, τα οποία μπορούν να διευκολύνουν την, σε ό,τι αφορά την ποιότητα της εργασίας. Και υπάρχουν πολλές διαφορετικές ερμηνείες. Άρα, για να υπάρχει μια κοινή βάση και να μπορούν να γίνουν συγκρίσεις μεταξύ των ταμείων, πήραμε τον ορισμό της ποιότητας ε, εργασίας της Eurofund και τα τέσσερα Eurofound και τα τέσσερα. Τονίζουμε δηλαδή την ε, εγγενή ποιότητα της εργασίας, οι ικανότητες που χρησιμοποιούνται, το κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον και η ένταση εργασίας και τέλος ποιότητα του εργασίας. Αυτό που σημειώνουμε φυσικά είναι ότι καμία δουλειά δεν τα πηγαίνει καλά και στις τέσσερις αυτές πτυχές και υπάρχουν ε, κάποιες υποχωρήσεις που θα πρέπει να κάνουν, για παράδειγμα οι θέσεις εργασία ε, που έχουν μεγάλα έσοδα συνεπάγονται και για να δούμε μια σύντομη επισκόπηση των τεσσάρων αυτών ταμείων που εξετάζουμε. Και γιατί? Γιατί πρόκειται για επιλεγμένα ευρωπαϊκά ταμεία που έχουν σημαντικές διαφορές σε ό,τι αφορά τη στοχοθεσία τους και σε ό,τι αφορά τους δικαιούχους και τα άτομα που αλλά και σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση που παρέχουν. Οι πιο βασικές διαφορές είναι ουσιαστικά μεταξύ του ορίζοντα 2020 και των τριών ε, υπόλοιπων ταμείων. Και αυτό γιατί ο ορίζοντας 2020 εργάζεται πιο πολύ και δραστηριοποιείται πιο πολύ στην της απασχόλησης. Και έτσι γίνονται λοιπόν συγκρίσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και του Ορίζοντα 2020, γιατί έχουμε πιο συγκρίσιμα, συγκρίσιμους τομείς εφαρμογής, αλλά αυτά που τελικά μοιάζουν είναι τον τρόπο με τον οποίο να διαπιστώνουμε ότι τα ευρωπαϊκά ταμεία μπορούν να υποστηρίξουν τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και την ποιότητα της εργασίας με διάφορους τρόπους κοιτάξαμε και τις νομοθετικές πράξεις από τις οποίες προέκυψαν τα ταμεία αυτά, γιατί δεν μπορούν φυσικά να ξεπεράσουν αυτά τα θέσεων απασχόλησης και στη διατήρηση των θέσεων αυτών απασχόλησης, κυρίως στις επιχειρήσεις και στους ακαδημαϊκούς κύκλους. Τα τρία υπόλοιπα ταμεία, το Ευρωπαϊκό και το Κοινωνικό Ταμείο, η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Απασχολησιμότητα των Νέων και το Ευρωπαϊκό Ταμείο για την Παγκοσμιοποίηση, προωθούν, αυξήσουν τι δυνατότητέ του για την αύρεση θέση απασχόληση. Να είναι πιο εύκολο δηλαδή να ενταχθούν στην αγορά εργασία τελικά τα άτομα αυτά. Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων είναι ουσιαστικά με ένα αντίτυπο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου με τη διαφορά ότι βάσει τη παγκοσμιοποίηση προσανατολίζεται στην επανένταξη σε μια βιώσιμη θέση εργασίας. Να πούμε για τα τρία αυτά μία. Το ενδιαφέρον είναι να κοιτάξουμε κατά πόσον οι θέσεις απασχόλησης που υποστηρίζουν είναι δευτερεύουσες. Υπάρχουν λοιπόν πολλές διαφορές ε, σε ό,τι αφορά τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης με τα διάφορα ευρωπαϊκά κονδύλια. Στον ορίζοντο 2020 και οι προκάτοχοι του προγράμματος έχουν δημιουργήσει πολλές θέσεις απασχόλησης, ιδιαίτερα στον τομέα αφορά την απασχόληση. Βρήκαμε φυσικά κάποια παραδείγματα. Και υπολογίζεται ότι ο ορίζοντας 2020 αναμένεται στην περίοδο 2014 και 2030 να υποστηρίξει 2,3 εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης. Οδηγεί τον κόσμο σε θέσεις απασχόλησης, αλλά 803.776 άτομα ήταν ήδη στην αγορά εργασίας όταν ξεκίνησαν στο πρόγραμμα. Και μετά από έξι μήνες, του Νορίου το 2020 βασίζονται σε οικονομικά μοντέλα, ενώ τα στοιχεία για τα τρία ταμεία προέρχονται από την υποβολή αναφορών των κρατών μελών. Να κοιτάξουμε το θέμα της ποιότητας, που είναι πολύ ενδιαφέρον. Τα απορίσματα είναι προοπτικές ε, σταδιοδρομία των ε, ερευνητών. Δεν έχουμε επαρκή στοιχεία σε ό,τι αφορά το ευρωπαϊκό επίπεδο για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, αλλά υπάρχουν στοιχεία σε επίπεδο κρατών μελών. Θα δώσουμε κάποια παραδείγματα. Το πιο ενδιαφέρον εργαλείο να μας ε, δώσει τις πιο πολλές πληροφορίες για την ποιότητα της απασχόλησης. Όχι όμως ακόμα και αυτό γιατί όταν δημιουργήθηκε η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων, υπάρχει, δημιουργήθηκε και υποχρέ, λοιπόν, προπόθεση. Αναμένουμε λοιπόν πιο πολλά στοιχεία, τα οποία όμως δεν έχουμε ακόμα στη διάθεσή μα. Το Ταμείο παγκοσμιοποίηση. Εδώ κοιτάξαμε και πάλι τις προοπτικές διαδρομίας και τι αντιλήψει των δικαιούχων για την ε, νέα θέση που έλαβαν. Αλλά και πάλι δεν έχουμε πάρει 20 καταδεικνύουν ότι εδώ υπάρχει βελτίωση της ε, μακροπρόθεσμης ασφάλειας για τη θέση απασχόλησης, ε, σταδιοδρομία, ε, αμοιβή των ερευνητών για τα άτομα που συμμετείχαν στις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και που βρήκαν θέση απασχόλησης. Βρήκαμε λοιπόν μεγάλη απόκληση στην ποιότητα της εργασίας και σε πολλές περιπτώσεις χαμηλή ποιότητα. Αλλά μπορούμε να εξετάσουμε και διάφορες πτυχές της ποιότητας. Και εδώ βλέπουμε ότι οι πιο πολλές ε, συμβάσεις ε, δεν είναι μόνιμες. Είναι ορισμένου χρόνου το εισόδημα των ατόμων αυτών ήταν αρκετά χαμηλό οριακά υψηλότερο από τον γιατί υπήρξε δουλειά, για παράδειγμα, σε βάρδιες, το οποίο δεν θεωρείται ιδανικό περιβάλλον για την εργασία. Παρ' όλα αυτά, 89% των ερωτηθέντων που συμμετείχαν στη μελέτη αυτή δήλωσαν ικανοποιημένοι γενικά με τις που συμμετείχαν στις έρευνες μας συμμετείχε στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και συμμετείχε μετά σε μία έρευνα για το τι έγινε για το μισθό του. Πολύ χαμηλό στην προκειμένη περίπτωση. Οι εργασιακές συνθήκες, οι οποίες όσα είναι ότι αυτή η δουλειά του είχε αλλάξει τη ζωή και ήταν ό,τι καλύτερο του είχε συμβεί. Είναι μόνο μία ιστορία φυσική, αυτή, μία μόνο περίπτωση περιπτώσεις όταν μιλάμε για την ποιότητα της εργασίας να έχουμε υπόψη μας ότι πρόκειται για ε, έναν όρο σχετικό και ότι αυτό που ε, και τη χορήγει στον κονδυλίο έχουμε διάφορες μεθοδολογίες σε ό,τι αφορά το θέμα. Δίνουν, δίνει συγκεκριμένες πτυχές και συγκεκριμένες ε, εκφάνσεις της ποιότητα της εργασίας. Δείκτε οι οποίοι περιλαμβάνουν πολύ πιο συγκεκριμένε και περιορισμένε παρατηρήσεις για την θέση απασχόληση. Έχουμε λοιπόν συμπεράσματα και συστάσεις και εδώ εστιάζουμε σε κάποια από τα βασικά σημεία. Αυτό που βρίσκουμε είναι πως η ποιότητα θα μπορούσε σε έναν ε, ε, καταστατικό κανονισμό να περιγράφεται καλύτερα. Αλλά βέβαια αυτό έχει θετικά και αρνητικά και υπάρχουν και εναλλακτικέ λύσεις που εξαρτώνται από το βαθμό φιλοδοξίας ε, που έχει τρίνουμε όσους εφαρμόζουν τα προγράμματα ή τα ταμεία να εξετάζουν και την πτυχή αυτή. Αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει ένα βασικό βήμα που ουσιαστικά είναι η σημερινή κατάσταση. Το επόμενο βήμα θα ήταν όχι μόνο να τονίζουμε τη σημασία αυτής τη ποιότητα, αλλά να τη στηρίζουμε με ενδεχομένως κατευθυντήριες γραμμές συστάσει που δεν είναι θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τις μελλοντικέ μελέτες και για τη μελλοντική εξέταση του θέματος της ποιοτική απασχόλησης. Και τέλος, στο υψηλότερο επίπεδο που θα ήταν μια αύξηση των ε, απαιτήσεων θα είναι κάτι αντίστοιχο με αυτό που έχουν θέσει απασχόλησης και βεβαίως τα στοιχεία αυτά να τα αναφέρουμε κατόπιν ε, προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τώρα, ε, έχουμε μια ερώτηση που πραγματικά είναι σημαντική, δηλαδή θα πρέπει όλα τα ευρωπαϊκά ταμεία να δημιουργούν και να στηρίζουν θέσεις απασχόλησης ή θα πρέπει οι συνέργειες μεταξύ των διαφόρων ταμείων και προγραμμάτων να την χάνουν καλύτερης χρήσης και εκμετάλλευσης. Γιατί το λέω, γιατί επειδή έχουμε αυτό το μοντέλο των ταμείων και το οποίο βρίσκεται κάτω-κάτω και μάλλον δεν το βλέπετε, αλλά αν το δείτε μέσα στην έκθεση θα το διαβάσετε πιο εύκολα, μας οδηγούν στο εξή συμπέρασμα, ότι αυτό που έχουμε στο αριστερό κομμάτι της εικόνας είναι το πιο σημαντικό, δηλαδή έχουμε την προσφορά και το εργαλείο που προσπαθεί να ενισχύσει την αγορά εργασίας και το εργατικό δυναμικό έτσι ώστε και η προσφορά και η ζήτηση μέσω των αντιστοίχων εργαλείων να ε, συνδυάζονται καλύτερα για να δημιουργούν νέες θέσει απασχόληση για όσου ήδη είναι στην αγορά εργασίας. Κάτι το οποίο θα βοηθούσε θα ήταν να είμαστε περισσότερο συνεπεί, τη στιγμή της μέτρησης τη ποιότητα ε, εγκάρσια στα ευρωπαϊκά ταμεία και εγώ βέβαια σκέφτομαι ως ερευνητής, αλλά γνωρίζω πως γίνονται προσπάθειες και σε διάφορα βήματα αλλά και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έτσι ώστε οι πληροφορίε να είναι πιο συνεκτικές, να υπάρχει καλύτερη συγκρισιμότητα μεταξύ ταμείων και ξέρουμε πόσες προσπάθειες κάνει και τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θεωρούμε πως υπάρχει ακόμα χώρος για βελτίωση στο κομμάτι αυτό και χρειαζόμαστε περισσότερα τεκμήρια για το πώς επηρεάζουν αυτές τις πολιτικές απασχόλησης τα ευρωπαϊκά ταμεία και κυρίως ποιες είναι οι μεθοδολογίες μέτρησης των επιπτώσεων έτσι ώστε να μετρήσουμε τις συνέπειες αυτές ανά μέσο. Και αυτό σε σύγκριση με άλλους παράγοντες που μπορεί να επηρεάζουν. Έτσι ώστε να έχουμε πιο πιστικά στοιχεία για το τι συμβαίνει τη στιγμή της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης ποιοτικών. Έχετε ερωτήσεις? Με μεγάλη χαρά να σας απαντήσω. Κάτι άλλο δεν έχω να προσθέσω. Σας ευχαριστώ πολύ. Η αλήθεια είναι πως έχετε πάρα πολλές ιδέες και καινοτομίες θα έλεγα μέσα στην έκθεσή σας και κυρίως μεταξύ αυτής της σχέσης η οποία δεν έχει την απαραίτητη συνέργεια μεταξύ ταμείων και η οποία θα μας βοηθούσε πολύ. Ε, κάποιος συνάδελφος... Α, ο κύριος ναι. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε. Έχω. Πιστεύετε ότι θα δημιουργούνταν αυτές τις θέσεις εργασίας αν υπήρχε λιγότερη γραφειοκρατική επιβάρυνση για τις επιχειρήσεις και κυρίως τις μικρομεσαίες στην ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Είπατε ότι κάνατε συνεντεύξεις, ότι είχατε ερωτηματολόγια. Τι ερωτήσει περιείχαν αυτά του προπολογισμού. Χρειαζόμαστε αποδείξεις. Άλλωστε το όνομά μου είναι και Θωμάς. Ο Θωμάς απαιτεί πιστήρια. Δεν ήταν ε, ικανοποιημένοι. Επομένως, σε τι πράγμα ακριβώ ήταν ικανοποιημένοι για να καταλάβω. Τα ταμεία και επιχειρηματική δραστηριότητα. Μπορείτε να μας δώσετε κάποιες λεπτομέρειες λοιπόν. Και επίσης μια ακόμη ερώτηση. Τι συγκεκριμένα θα μπορούσε η διασύνδεση με τα ταμεία και τις δράσεις αυτές. Θα ήθελα απλώ να σας ευχαριστήσω για την παρουσίαση που κάνατε και είναι κάτι που είπατε που πραγματικά με εντυπωσίασε. Σε απασχόλησε αυτό είναι ουσιαστικό. Αυτό που μας ενδιαφέρει πάντα είναι τη στιγμή της εφαρμογής του ελέγχου των προϋπολογισμών. Πώς μπορούμε να αξιολογούμε αυτά τα αποτελέσματα, γιατί πολλές φορές εμείς λαμβάνουμε μόνο αριθμητικά στοιχεία. Και είναι ενδεχομένω τα αποτελέσματα. Στην αρχή της παρουσίασης είπατε πως ένα από τα θετικά του Horizon 2020 είναι η προσέγγιση που ακολουθεί που είναι ότι βασίζεται στην ζήτηση ενώ τα υπόλοιπα είπατε ε, πω η καλύτερη λύση ή μία από τι λύσει θα ήταν να προσπαθήσουμε να έχουμε προγράμματα στα οποία θα ισορροπήσουμε μεταξύ προσφοράς και ζήτησης έτσι ώστε να έχουμε μια πιο ισορροπημένη δυναμική και όχι μόνο προσφορά γιατί αυτό πολλές φορές καταλήγει σε σας ευχαριστώ πολύ για τα ερωτήματά σας που ήταν πολλά. Δεν θα ακολουθήσω την ίδια σειρά στις απαντήσεις μου, αλλά θα προσπαθήσω να τα απαντήσω όλα. Μεθοδολογία. Είναι πολύ σημαντική ερώτηση και όντως δεν στάθηκα αρκετά. Πριν εξηγήσω τη μεθοδολογία, ίσως πρέπει να επαναλάβω ποιος ο στόχος της μελέτης. Ίσως εκεί να υπάρχει κάποια παρανόηση. Μας ζητήθηκε να συγκρίνουμε τέσσερα ταμεία, τα οποία είχατε επιλέξει εσείς και τα οποία περιγράφονται, για να δούμε τι στοιχεία υπάρχουν ε, σχετικά με τα αποτελέσματα αυτών των ταμείων σε επίπεδο θέσεων απασχόλησης και ποιότητας αυτής της απασχόλησης. Δεν μας ζητήθηκε να αξιολογήσουμε ευρύτερα το, τις επιπτώσεις των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Αυτό ξεπερνά το πεδίο εφαρμογή της μελέτης μας. Εμείς ουσιαστικά κάναμε μία προσπάθεια περιγραφής των αποτελεσμάτων που βρίσκουμε, συλλέγοντας όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία και δίνοντας μια αφετηρία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να συζητήσει το θέμα της ε, δημιουργίας θέσεων εργασίας και κυρίως των θέσουν εργασίες υψηλής ποιότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μεθοδολογικά βασιστήκαμε σε ποιοτική έρευνα με δύο διαφορετικές αξιολογήσεις ε, εγγράφων. Πρώτα απ' όλα εξετάσαμε τα έγγραφα που σχετίζονται με τα ευρωπαϊκά ταμεία, δηλαδή τους κανονισμούς χρηματοδότησης των τεσσάρων και επίσης όλες οι επιπτωσιολογικές μελέτες που ήταν διαθέσιμες, όπως επίσης και οποιαδήποτε αξιολόγηση αυτών των ταμείων και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και σε εθνικό επίπεδο. Σε εθνικό επίπεδο για τα διαστροτικά ταμείο και πάλι εδώ είναι πολύ ευρύτερα οι συνέπειες από αυτές που έχουμε στο πεδίο εφαρμογής μελέτης μας και θα έπρεπε να κάνουμε ε, μία συλλογή των όσων στοιχείων έχουν σε περιφερειακό επίπεδο τα κράτη-μέλη, οπότε εμείς κοιτάξαμε μόνο έναν επιλεγμένο αριθμό κρατών μελών, όπου θεωρήσαμε ότι μπορεί να έχουμε αποτελέσματα και για την αριθμό θέσεων απασχόλησης και για την ποιότητα αυτών των θέσεων. Να μετρήσουμε ε, πιο συγκεκριμένο το θέμα της ποιότητας της θέσης απασχόλησης αλλά και τον αριθμό των θέσεων απασχόλησης ακολουθώντας τους δείκτες εύξης με αρκετούς εμπλεκόμενους σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και σε εθνικό επίπεδο. Και εξετάσαμε και τον αριθμό παράδειγμα θέσεων απασχόλησης που δημιουργήθηκαν. Εμείς δεν είχαμε σκοπό να μετρήσουμε τις επιπτώσεις των ε, χρηματικών, ε, χρηματοδοτικών αυτών εργαλείων στα κράτη-μέλη. Δεν ήταν η μελέτη ε, αυτή. Και την ερώτησή σας, δηλαδή το αν θα μπορούσαν να έχουν δημιουργηθεί από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία πιο ποιοτικέ θέσεις εργασίας και αν το διοικητικό βάρος ή οι εφαρμοστικές δυσκολίες επηρέασαν, να σας πω πως δεν γνωρίζω δεν έχουμε στοιχεία σχετικά σε εθνικό επίπεδο για να συγκρίνουμε με το ευρωπαϊκό επίπεδο. Φαντάζομαι ότι χωρίς την παρέμβαση των ευρωπαϊκών κονδυλίων θα ήταν δύσκολο. Αλλά αυτό ακριβώς είναι και η δική μας σύσταση, να γίνει κάτι τέτοιο γιατί εμείς είμαστε περισσότερο, ε, παροτρύνουμε μάλλον γίνουν περισσότερες επιπτωσιολογικές μελέτες για το τι θα είχε συμβεί αν δεν είχαν, τα, αν δεν είχαν παρέμβει τα ευρωπαϊκά ταμεία. Ε, παροτρύνουμε μάλλον γίνουν περισσότερες επιπτωσιολογικές μελέτες για το τι θα είχε συμβεί αν δεν είχαν, τα, αν δεν είχαν παρέμβει τα ευρωπαϊκά ταμεία. Θα είχαν δημιουργηθεί παρόλα αυτά αυτέ οι θέσει απασχόληση. Έχουμε κάποιες μελέτες και σε ευρωπαϊκό επίπεδο που έχει ζητήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κάποιες που έχει ζητήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και επίσης γίνονται τέτοιες μελέτες και σε εθνικό και σε περιφερειακό επίπεδο, οπότε κάποια στοιχεία. Για τη δεύτερη ερώτηση, ρωτήσατε αν η δημιουργία θέσεων απασχόλησης εξαρτώνται από τις εξελίξεις στην οικονομία ή αν εξαρτώνται από την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Μα νομίζω ότι αυτό... Τι είδου τεκμήρια και αποδείξει έχουμε. Νομίζω ότι θα βρείτε κάποια από αυτά στην έκθεση. Έχουμε δώσει και κάποια παραδείγματα και θα σας έλεγα να τα διαβάσετε. Προκύπτουν ήδη από τις ευρωπαϊκές μελέτες είτε από τις εθνικές μελέτες. Σας παρακαλώ πολύ να λάβετε υπόψη ότι από τις οκτώ κρατημέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να κάνουμε μια προσπάθεια απογραφής για το τι είναι διαθέσιμο. Εμείς δεν μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό σε βάθος. Κάτι τέτοιο θα ήταν πολύ χρήσιμο και ίσως μια ευκαιρία ε, για μας. Ίσως το σκέφτεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή τη στιγμή στα πλαίσια του. Σε ερώτηση για τα αριθμητικά στοιχεία που έδωσα στην παρουσίαση. Νομίζω ότι μιλήσατε για το 89% που είναι ακόμα ικανοποιημένοι και είπατε από πού προκύπτει αυτό το νούμερο. Και γιατί δηλώνουν ικανοποίηση. Ο αριθμός μια καλή μελέτη με ένα δείγμα 2.000 ε, συμμετεχόντων ήταν στοχευμένο και τυχαίο δείγμα ε, δικαιούχων από το ΕΚΤ. Κάποιοι βρήκαν δουλειά, κάποιοι όχι. Και στην... Ε, στο επίπεδο ικανοποίησης νομίζω πάντως είναι έτσι όπως τα είχαμε πει. για τις συνέργειες μεταξύ των ταμείων και εδώ θα πρέπει να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, νομίζω ότι έχετε το δίκιο. Πολύ καλή παρατήρηση. Ε, σύγκριση μεταξύ τόσο διαφορετικών ταμείων, γιατί το Horizon 2020 με το ΕΚΤ. Μπορούμε να το συστήσουμε, γιατί για εμάς κάποια άλλα ταμεία ή εργαλεία θα ήταν πολύ καλύτερα ε, για να κάνουμε μια σύγκριση της ομάδας υψηλού επίπεδου για το Horizon 2020 και τα μελλοντικά προγράμματα πλαίσιο για τις ιστορίες να μην έρχονται αρκετά κοντά στον πολίτη. Όταν κάνει κανείς ε, ε βασική έρευνα, δύσκολο πλησιάζει το πολίτη. Συμβαίνει ε, η πολύ σωστή, ακριβή δική μας δουλειά επισκιάζεται από όχι τόσο ακριβής. Εδώ ή αν στο μακροοικονομικό, χωρίς να ενοχλούμε τόσο πολύ τις επιμέρους επιχειρήσεις, μπορούμε να έχουμε επαρκή στοιχεία. Ε, σε αυτό θα... Ευχαριστώ πολύ για την έκθεση λοιπόν, θα την αξιοποιήσουμε για τις συνεργασίες ε, πιο πολύ. Αλλά πρέπει να συμμετέχουν και τα κράτη-μέλη, τοπικές αρχές και το καθεξής. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Έχετε εσείς το λόγο τώρα. Madame Grisard, je suis la directrice d'investissement de la DG Emploi. Grisard, διευθύντρια από τη Γενική Διεύθυνση για την Απασχόληση, προσωρινή. Έχουμε λοιπόν προχωρήσει στις αναλύσεις που θα σας ετοιμάσουμε για το τέλος του μήνα και για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Προσπαθούμε να βελτιώσουμε τη συνεργασία με τα προγράμματά μας, μέσα στα προγράμματά μας που θα συγχωνευτούν μεταξύ τους, όχι όμως με τον όριο 2020, γιατί είναι τελείως διαφορετικές οι αποστολές μας. Λαμβάνουμε υπόψη ε, τη μελέτη, συμμεριζόμαστε πολλά από τα συμπερασματά τη. Η ποιότητα των θέσεων εργασία όντω είναι δύσκολη να εξασφαλιστεί. Σειρά δικτών που αντικατοπτρίζουν και τι διαφορέ μεταξύ των πρώτων μερών αλλά και τι διαφορέ μεταξύ των διαφορών δράσεων και από τη τελευταία μελέτη που δημοσιεύσαμε για τις θέσει που, για, ε, για τα επαγγέλματα που έχουν ε, παρουσιάζουν ελληματική εικόνα και άλλα που έχουν πλεονασματική. Στην ελληματική εικόνα μπορεί να είναι ε, θέσει εργασίας και μακροπρόθεσμης ακόμη και με καλής αμοιβή, ε, αλλά και χωρίς υψηλή κατάρτιση όπως ε, στην, στον κατασκευαστικό κλάδο αλλά βέβαια και στον ιατρικό κλάδο. Υπάρχουν πολλές δηλαδή διαφορετικές κατηγορίες επαγγελμάτων που λείπουν. Άρα, εάν η δράση των κονδυλίων περιοριστεί σε πολύ συγκεκριμένο βαθμό στην ποιότητα της απασχόλησης, θα είναι δύσκολο να βρούμε θέσει εργασία για εκείνου στου οποίου ουσιαστικά υπευθύνει τη δουλειά μα, δηλαδή αυτού που δυσκολεύονται περισσότερο να βρούμε θέση εργασία. Ε, ξέφρασε την απορία του για το επίπεδο ικανοποίηση. Μα φυσικά αν ταλαιπωρηθεί κανεί τόσο πολύ μέχρι να βρει μια θέση απασχόληση, την ώρα που θα τη βρει θα είναι πολύ ικανοποιημένο. Και α μην είναι η ιδεώδη θέση εργασία. Όταν κανεί ψάχνει για ένα χρόνο και βρει τελικά κάτι, είναι ικανοποιημένο. Η έκθεση επίσης μας δείχνει ότι τα τρία ταμεία ε, στόχο έχουν την επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο, όχι στη δημιουργία θέσης εργασίας. Είναι η αντίστροφη δηλαδή προσέγγιση. Εμείς βελτιώνουμε την απασχολησιμότητα εκείνων που δυσκολεύονται και δι, ε, εκείνων που δυσκολεύονται περισσότερο από τους άλλους να βρουν μια θέση εργασίας. Ως ε, μέλος και εγώ του, ερευνητικού κόσμου του, ερευνητικού έχω και εγώ σαν τον Άγιο Θωμά την ε, απέτηση να βλέπω αποδείξεις ήμουνα μάλιστα και δημοσιονομικής ελεγκτής στο παρελθόν ε, είναι βέβαια ε, απαραίτητο να σας καταστήσω σαφές ότι αυτές οι εκτιμήσεις και αξιολογήσεις που υπάρχουν σε μεγάλο βαθμό κοστίζουν πολύ και όπως είπαν και οι συνάδελφοι από την άλλη Γενική Διευθύνση δεν είναι πάντα πρόθυμοι οι αποδέκτες των αξιολογήσεων των πληροφορίες. Και επίσης ε, έχουμε να κάνουμε και με αξιολογήσεις οι οποίες μερικές φορές ακολουθούν, για να εξηγήσω τους όρους, την μεθοδολογία της ιατρικής. Όταν δηλαδή η ιατρική δοκιμάζει ένα φάρμακο με παράλληλη χρήση του πλασέμπο. Στο μισό πληθυσμό δίνει το φάρμακο και στον άλλο μισό το πλασέμπο. Εάν όμως εγώ πάω στην κατερπίλαρ και πω σας δίνω 15 ε, θέσεις εργασίας πραγματικές και άλλες 15 που θα είναι πλασέμπο, ε, τότε δεν πρόκειται να με ε, ακούσουν. Άρα βεβαίως ναι πρέπει πάντα να γίνονται μελέτες με αντιπαραβολή βεβαίως. Και να ενημέρωσες τα συζητήσαμε, περιμένουμε περισσότερες πληροφορίες από τα κρατη πριν να κλείσει ο χρόνος για να αντιληφθούμε καλύτερα την αποτελεσματικότητα του ΓΕΙ σε φυσιολογικούς όρους και επίσης βελτιώνοντας τους δείκτες ε, ποιότητας στην παρακολούθηση της δράσης ε, και για τους νέους μετά ε, εξάμηνο, 18 δεκαοκτάμηνο από την εξέβριση της εργασίας ε, κοιτάμε πάντα να δούμε πού βρίσκονται για να αξιολογήσουμε τα προγράμματα. Μήπως κάποιος από τους συναδέλφους θέλουν να ρωτήσουν κάτι ακόμα. Νομίζω πως η μελέτη έχει πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία και θα τα κοιτάξουμε σε βάθος και νομίζω ότι είναι φυσιολογικό αυτό που μας απάντησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Περιμένουμε να δούμε τα νέα προγράμματα έτσι ώστε ε, να διαπιστώσουμε πώς τα, οι πρακτικές από κάποιο κλάδο θα, ή κάποιο, κάποιο ταμείο θα μπορούσαν να εφαρμοστούν και στα υπόλοιπα. Γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε κάποια άποψη η οποία επηρεάζεται και από τις πληροφορίες που φτάνουν μέχρι εμάς. αυτή τη στιγμή από γράμματα πολύ μεγάλα δεν έχουν την ίδια φήμη. Και δεν μιλώ μόνο για την απασχόληση, που είναι και το βασικό που μας ενδιαφέρει, αλλά και άλλες διαστάσεις που υπάρχουν. Ίσως θα μπορούσαμε να ακολουθήσουμε την ίδια φόρμουλα και να δούμε τι γίνεται ε, τα όσα βγάζει ένα σταζιέρ στο Horizon 2020 ε, είναι ένα καλό ποσό, θεωρείται πετυχημένο ή πετυχημένα. και δεν θεωρούνται ως επένδυση στο μέλλον από ανθρώπους που βρίσκονται σε κλάδους που έχουν μεγάλο πρόβλημα απασχόλησης. Δεν μιλώ για το κατά πόσο κάποιος είναι. Νομίζω πως μας δώσατε πάρα πολύ τροφή για σκέψη. Θα τα κοιτάξουμε σε βάθος και θα κάνουμε τη συζήτηση για το πώς θα εφαρμόσουμε όλες αυτές τις ε, μελέτες στον καινούριο προϋπολογισμό, έτσι ώστε να βελτιώσουμε τις επιδόσεις μας. Αν δεν υπάρχουν λοιπόν, ευχαριστώ που ήρθατε. Δίνω το λόγο τώρα στον ε, συνάδελφο κύριο Σαρβαμά τη θέση εδώ στο Προεδρείο γιατί ε, ε, έχω και κάποιες άλλες συνεδριά στο πρόγραμμα και θα αναλάβει την Προεδρία για το υπόλοιπο της... Καλησπέρα και από μένα. Χαίρομαι που ε, την εσύ απαλλαγής ε, για το έτος 2017 για τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς το Μιρμάρ Βερμανία και θα δώσω το λόγο κατευθείαν στην κυρία Μπετίνα Γιάκοψ, στην εκπρόσωπο του Ευρωπαϊκού σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να σας παρουσιάσω την ειδική έκθεση για την, Ευρωπαϊκή, για την συνδρομή ε, της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης προς τη Μιερμάρ Βερμανία. Βρίσκεται σε μεταβατική ε, φάση από τον Μάρτιο του 2011. Ο πληθυσμό είναι αποτελείται από πολλέ εθνικέ ομάδε, οι οποίε σε διάφορε περιστάσει και διάφορε ιστορικέ στιγμέ έχουν ε, αποδεθεί σε πολέμους, συγκρούσεις, ε, διατρησκευτικούς, διαθνοδικούς και οι κυρώσεις που είχαν εφαρμοστεί στην κυβέρνηση τον Απρίλιο του 2012 έχουν ανασταλεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι το 2013. Όλες οι κυρώσεις λοιπόν είχαν ανασταλεί εκτός από το εμπάργκο όπλων. Πάνω από ένα δις ε, έχει δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την περίοδο 2007 μέχρι 2020 μέσω θεματικών διμερών εργαλείων κυρίως άμεσες και έμεσες λοιπόν επιδοτήσεις, ε, παροχές ε, κονδύλια. Επικεντρωνόμαστε στα εργαλεία του 2012-2016 μέσω του εργαλείου α, συνεργασίας. Δεν καλύπτουμε δηλαδή το νέο κύμα βίας κατά, ε, κατά το Ροχίνγκα. Ποιες ερωτήσεις λοιπόν θέσαμε κατά τη διάρκεια της έρευνας. Θέλαμε βασικά να διαπιστώσουμε κατά πόσο η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Μιανμάρ ήταν αποτελεσματική. Έγινε από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είχε θέσει συγκεκριμένες ε, προτεραιότητες. Εκτιμήθηκε επίσης η τη Ευρωπαϊκή Αναπτυξιακή Βοήθειας και αναρωτηθήκαμε κατά πόσο έχουμε πετύχει τους στόχου μα. Ποια ήταν λοιπόν τα πορίσματά μας. Η έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η αναπτυξιακή βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν μερικώ αποτελεσματική. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έπαιξε σημαντικό ηγετικό ρόλο στην πρόθεση των προτεραιοτήτων ανάπτυξη και χορήγησε σημαντική χρηματοδότηση προς τη χώρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανταποκρίθηκε ενεργά στις ανάγκες της χώρας σε δύσκολες ε, στιγμές, όπου το θεσμικό σύστημα και η βούληση και η ταχύτητα των μεταρρυθμίσεων ήταν ε, επισφαλής. Εκτιμήθηκαν λοιπόν οι ανάγκες και η επιλογή των ε, προτεραιοτήτων δεν ήταν αρκετά στοχευμένη. Διαπιστώσαμε ότι η πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή να, να εντοπιστεί σε τέσσερι τομεί δεν συνάδουν με την ατζέντα του 2012 για αλλαγή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίση δεν εκτίμησε επαρκώ τι γεωγραφικέ προτεραιότητε στο εσωτερικό τη χώρα. Η κινητοποίηση του εγχώριου, των εγχώριων κονδυλίων δεν ε, συμπεριληφθήκε στι βασικέ προτεραιότητε παρά το γεγονό ότι αποτελεί βασικό παράγοντα για την ανάπτυξη τη χώρα. Επίση, η διαχείριση τη αναπτυξιακή βοήθεια ήταν γενικώ πω ικανοποιητική. Οι ενέργειε στράφηκαν προ τι προτεραιότητε τη ανάπτυξη για ανάπτυξη ε, της χώρας και η επιλογή οκτώ τρόπων παροχή βοήθειας ήταν σωστή. Ωστόσο, η αιτιολόγηση του ποσού που ταπανήθηκε σε κάθε τομέα δεν ήταν καν Στην περίοδο 2012-2016 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, χρησιμοποίησε τους όρους αντιμετώπισης κρίσεων για να έρθει σε άμεση επαφή με τους ε, ομολόγους μας. Αυτό μείωσε τη διαφάνεια της διαδικασίας και μείωσε την απόδοση των κονδυλίων σε ό,τι αφορά το έργο. Τώρα, το ποσοστό επιτυχίας των έργων ήταν ε, διαφορετικό. Υπήρξαν σε κάποιες περιπτώσεις καθυστερήσεις και αυτές οι καθυστερήσεις σήμαιναν ότι δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε τη βιωσιμότητα των πόρων για το ίμιση σχεδόν των έργων. Τι προτείνουμε. Είναι Επομένως, είναι απαράδεκτο να πρέπει να φτάσουμε το Σεπτέμβριο του 2016 για να γίνει μια πρώτη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των δύο γενικών διευθύνσεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πιστεύω θα έπρεπε να έχει θεσπίσει ένα κοινό σχέδιο για την ε, κατεπίγουσα αναπτυξιακή βοήθεια σε περιοχές πληττόμενες μακροπρόθεσμα από κρίση. Η κρίση των Ροχίνκα επίσης μας φέρει ενώπιον του εξής ακατανόητου γεγονότος. Πώς είναι δυνατόν να μην χορηγηθούν κονδύλια για την ειρήνη στο Ρανκίν και βλέπω ότι έχουμε χάσει, όπως λέει άλλωστε και το ελευθερικό συνέδριο, μια μεγάλη ευκαιρία για μια περιοχή που θα μπορούσαμε να έχουμε βοηθήσει μια περιοχή ιδιαίτερα ευάλωτη. Γι' αυτό παρακαλώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επεκτείνει το πεδίο εφαρμογή του Ταμείου αυτού και για το κράτος του Ρακίνα. Βεβαίως, οι ενισχύσεις προς την ε, Μιανμάρ Βυρμανία δεν μπορούν να αξιολογούνται μόνο υπό το φως της κρίσης των Ροχίνγκα και γι' αυτό θα ήθελα να επανέλθω σε κάποια συγκεκριμένα ε, σε κάποια πιο γενικά μάλλον σημεία της ε, ειδική έκθεση και τα πω ό,τι λέει το ελεγκτικό συνέδριο, δεν θεωρώ ότι θα έπρεπε να έχει περιοριστεί σε κάποιου συγκεκριμένου τομεί προτεραιότητα η ευρωπαϊκή βοήθεια. Κατάρτιση, διακυβέρνηση, διοίκηση, ειρήνη θα έπρεπε να είναι η τομή προτεραιότητα για τη χρηματοδότηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η μετάβαση στη συνέχεια σε δύο τομεί προτεραιότητα μόνο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάντως πιστεύω στο μέλλον θα πρέπει να αιτιολογεί καλύτερα τις επιλογές της στους τομεί χρηματοδότησης ως προς τις δράσεις και του τομεί προτεραιότητα. Και για να το επιτύχει αυτό θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να ενισχύσει τη συνεργασία της ε, με τους διεθνείς εταίρους στη Βυρμανία ώστε να βελτιώσει με οικονομίες κλίμακος τις δράσεις πολλαπλών χορηγών και να βελτιώσει τη διαχείριση των έργων που χρηματοδοτεί ώστε να λάβουν μεγαλύτερη ορατότητα η δράση που χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση Ένωση και τρίτον να εξασφαλίσει παρακολούθηση τις συνέχεια που δίνεται στις δράσεις και τα έργα. Αυτές είναι οι συστάσεις μου, αυτά είναι τα όσα σκοπεύω να περιλάβω στο έγγραφο εργασίας, το οποίο πρόκειται να δημοσιεύσω στις ε, προσεχείς εβδομάδες. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ κύριε ε, Πανιό και πολύ σύντομα θα ακούσουμε τους Κιώδης εισηγητές. Αν δεν περάσει κανείς ε, την... Ε, αν δεν διαβεί κανεί το κατόφλι της, αίθουσα αυτή, θα ακούσουμε τον κύριο Τσέλερ πρώτο και τελευταίο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον κύριο Παρνιού για την έκθεση και την ε, έκθεση που θα καταρτήσει. Βεβαίω δεν είναι εύκολο να περιγράψουμε μέσα σε λίγε λέξει μόνο την κατάσταση στη Μιανμάρ. Πριν από μερικέ εβδομάδε την επισκεφθήκαμε μια αντιπροσωπεία τη Υποεπιτροπή των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για να διαπιστώσουμε ότι η κατάσταση στη χώρα, όχι μόνο μάλιστα σε σχέση με του Ροχίνγκα και την έξοδο, την ε, εκδίωξή του προ τον Μπαγκλαντέ, αλλά και γενικότερα έχει επιδεινωθεί σημαντικά. Λαμβάνουμε δε τι τελευταίε ημέρε ε, από το Κατσίν, ε, το Βορρά, αλλά και γενικότερα από την Βυρμανία, οι ειδήσει που μας μιλούν για εθνοτικές ομάδες που πέφτουν θύματα των πολεμαρχών που προσπαθούν να επικυριαρχήσουν στις περιοχές αυτές και άρα γίνονται συγκρούσεις με πολύ άριθμους νεκρούς από ό,τι φαίνεται, πράγμα το οποίο ασφαλώς δεν βελτιώνει την κατάσταση στη χώρα. 2011-2012, ίσως και υπό την εντύπωση μιας εν μέρη προσπάθειας, μερικής προσπάθειας εκδημοκρατισμού και βέβαια με το βραβείο Ζαχάροφ και την εκλογή της Αντζουκή στη θέση του Προέδρου της χώρας ε, είχαμε ε, ένα κλίμα εφορίας ότι τα πράγματα πάνε καλύτερα και έτσι προσφέρθηκε μαζική υποστήριξη προς τη χώρα. Πάντως παραμένει η κατάσταση λίγο πολύ όπως την ξέραμε, εν μέρει έχει προχωρήσει ο εκδημοκρατισμός, σε ένα βαθμό εκπροσωπείται η κοινωνία των πολιτών μέσα από το κοινοβούλιο, ενώ σε μεγάλο βαθμό τον έλεγχο και των πόρων και της χώρας τον έχει ο στρατός. Δεν υπάρχει δηλαδή περίπτωση να εισαγάγει το Κοινοβούλιο νομοθεσία και να εγκριθεί αυτή χωρίς την έγκριση και επεξεργασία βέβαια από τον στρατό, ο οποίος λίγο πολύ ανήκει σε ένα στρατιωτικό βιομηχανικό σύμπλεγμα πάρα πολύ στενά δεμένο με την Κίνα και εδώ έχουμε άλλωστε να εντοπίσουμε και τα αδύναμα σημεία της πολιτικής της ε, ανάπτυξης που ακολουθούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι μέσω, ε, επειδή εργαζόμαστε μέσω διαφόρων καταπιστευμάτων και άλλων φορέων περιορίζεται η ορατότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πολλές φορές οι εταίροι Ε, συμμετέχουν σε αυτή τη δουλειά και κάνουν ένα μέρος της δουλειάς, χωρίς όμως να φαίνεται να είναι εξίσου αποτελεσματική όσο εμείς από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης θα απαιτούσαμε. Και βέβαια για την κοινωνία των πολιτών, για την Μιανμάρ ε, Βιρμανία ιδιαίτερος εξαίρει το ελεκτικό συνέδριο τη σημασία των ε, έργων μικροχρηματοδότησης, που έχουν ε, επιτρέψει σε πολίτες ε, να δραστηριοποιηθούν ή να σταθεροποιηθούν στον χώρο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ε, άλλο ζήτημα βέβαια χρήσιμο ήταν το άνοιγμα της ευρωπαϊκής αγοράς για την Βυρμανία που έφερε κάποιους καρπούς μέσα σε πολύ, λίγο, σε πολύ μικρό χρονικό, χρονικό διάστημα, εξασφαλίζοντα τη δημιουργία 150.000 θέσεων εργασία μόνο για τον χώρο της φαντουργίας. και είμαστε πεπισμένοι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη πρέπει να μεριμνούν να τηρούνται πάντοτε οι όροι οι κοινωνικοί όροι και οι εργασιακές σχέσεις που απαιτούνται στις θέσεις αυτές εργασίας επεσήμανε ο συνάδελφος Παρνιό ότι θα περιγράψει την κατάσταση σε μια πληρέστερη ε, έκθεση και μάλιστα όχι μόνο για την ε, Μιανμάρ αλλά και για τη γενικότερη αναπτυξιακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ευρύτερη περιοχή. Νομίζω ότι θα πρέπει να διατυπώσουμε τις επικρίσεις μας σε σχέση με το θέμα αυτό μέσα από την έκθεση. Σας ευχαριστώ πολύ και θα δώσω τώρα το λόγο στην Γενική Διεύθυνση ΔΕΦΚΟ πριν ακολουθήσουν οι επόμενοι ομιλητές. Σας παρακαλώ. Εγώ είμαι σκιώδης όμως, θα ήθελα να μιλήσω. Δεν έχω λάβει αυτές την... Συγγνώμη, δεν ενημερώθηκα. Ε, παρακαλώ, προχωρήστε. Άντε να τα πω και εγώ στα γερμανικά, μια και έχουμε τους διερμηνείς εδώ τρέφαμε ελπίδες ότι θα βελτιωθεί πραγματική κατάσταση και ότι η ε, επικυριαρχία του στρατού θα μπορούσε μέσα από μια διαδικασία εκδημοκρατισμού να περιοριστεί, πράγμα το οποίο σε πολύ περιορισμένο βαθμό μόνο Υλοποιήθηκε άλλωστε και η έκθεση επισημένη της ε, διαφορές στο ότι η κατάσταση ήταν αυτή που ήταν το 2013, άρα είναι κατανοητή η δέσμευση αυτού του δισεκατομμυρίου. Θέλαμε να υποστηρίξουμε τη διαδικασία του εκδημοκρατισμού, να μην υπάρχουν οπισθοδρομήσεις, να μην υπάρχουν ε, προβλήματα στην πορεία του εκδημοκρατισμού. Ο κύριος Παρνιό, ο κύριος Σέλερ μίλησαν έχει μια διατύπωση μάλλον προσεκτική, ας το πω έτσι, ενώ υπάρχουν κάποια σημεία στα οποία θα, θα μπορούσαν να είναι πολύ πιο ανοιχτή η διατύπωση της έκθεσης του λεκτικού συνεδρίου. Η κατάσταση έχει ριζικά αλλάξει, όπως άλλωστε ανέφερε και ο Ζιλ, με την εθνοκάθαρση των Ροχίνγκα. Ξεκινήσει με μέτρα αναπτυξιακά και ε, υποστήριξη θα έπρεπε να παραμείνει ως αν θα έπρεπε να τροποποιηθεί και ως προς τη γεωγραφική του, το γεωγραφικό του προσανατολισμό, αλλά και ως προς τις επιμέρους προτεραιότητες των έργων. Δεν τηρήθηκαν. Μεγάλες υποσχέσεις είχαν δοθεί ότι θα επιτραπεί επάνωδος από τον Μπαγκλαντές τον Ρογίνγκα, δεν έχει γίνει, τον δεν έχει γίνει τίποτα. Ούτε καν βέβαια θα είχαν μια ευκαιρία να γυρίσουν θα ήταν σκόπιμο να γίνει ένας επαναπροσδιορισμός ε, του προγράμματος. Και αυτό άλλωστε βλέπω ότι δεν το έχει διατυπώσει σαν πρόταση το ελεκτικό συνέδριο, που επιμέρους βλέπω να έχει κάποια σωστά σημεία και θα συμπληρώσει και ο Σίλ με τις δικές του παρατηρήσεις. Αλλά ε, θεωρώ... Ενθαρρύνω λοιπόν την Επιτροπή, εν πάση περιπτώσει της υποβάλλω το ερώτημα, εάν υπάρχει... Ευχαριστώ κύριε Κλίντ. Θα δώσω τώρα το λόγο στην Γενική Διεύθυνση ΤΕΦΚΟ. Σας ευχαριστώ πολύ. Έχουν υπογραφεί ήδη και δύο από αυτές είναι πανεθνικές. Εκεί βρισκόμαστε για τις συστάσεις του ελεγκτικού είναι να εστιάσουμε για να πετύχουμε αποτελέσματα. Μα ζητήθηκαν να στηρίξουμε τις εκλογές των εκτιμήσεων και τους δωρητές. Ίσως θα μπορούσαμε αυτά να τα έχουμε επισημοποιήσει περισσότερο. να θεωρηθεί ως πιλωτικό ε, το θέμα της ανθρωπιστικής ε, βοήθειας ε, στην Μιανμάρ και εδώ έχουμε επισημοποιήσει το θέμα αυτό με την εκπαίδευση για τις περιοχές όπου ζουν εθνικές μειονότητες σε συνεργασία με την ΕΚΟ και αυτή η επισημοποίηση Τώρα για την ε, στενότερη παρακολούθηση των παραδοτέων εμείς πάντα προσπαθούμε να μετρήσουμε τα αποτελέσματα και πάντα χρειάζονται αποτελέσματα. Είναι πολύ αδύναμες οι στατιστικές ε, που συλλέγουμε και έχουμε προσπαθήσει πάρα πολύ και δεν έχουμε αρκετή για να συλλέγει αυτή τα δικά της δεδομένα γιατί δεν μπορεί να χαράσει πολιτική μια κυβέρνηση χωρίς να ξέρει τι γίνεται εκεί που, υπάρχουν και περιοχές με πάρα πολλές εθνικές μειονότητες και είναι δύσκολο οι πληροφορίες αυτές να φτάσουν στο κέντρο. Πάντως και εκεί η παρακολούθηση ε, ισχυροποιείται και ε, χαίρομαι που λαμβάνουμε υπόψη και αυτή τη σύσταση για τη διαχείριση των project, για τις δράσεις μας και για το να είμαστε πιο ορατοί. Το προφίλ μας μέσω μιας, συγκεκριμέ... μιας ε, ενιαίας σύμβασης που θα προωθεί όλες τις ευρωπαϊκές δράσεις στη χώρα.